το θέμα αυτό το οποίο αφορά την διεθνή αυτή συμφωνία για το κέντρο τεχνολογίας και επιστήμης είχε ιδρυθεί το 1994 στην ε, Μόσχα και στόχο είχε ακριβώς να μην πέσει η τεχνολογία της έσοδου στα λάθος χέρια. Όμως εφόσον έχουν πλέον μειωθεί η εμπιστοσύνη και έχουν αποκλίνει οι πολιτικοί στόχοι η Ρωσική Ομοσπονδία το 2010 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ε, ε, συμφωνία αυτή, η οποία ετέθη ισχύ τον Ιούλιο πέρσι. Συνήθη μια νέα συμφωνία, ένα νέο κέντρο με έδρα την Αστάνα του Καζακστάν. Το Κοινοβούλιο συνεχίζει βεβαίως τις ε, επαφές το, η συμφωνία συνέχειας του Διεθνούς Κέντρου θα διασφαλίσει ότι τα υφιστάμενα και τα νέα έργα θα συνεχίσουν με τη νέα σύνθεση με ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο κάλυψης και με στόχους που αφορούν συγκεκριμένα την τεχνολογία διπλής χρήσης. Ο κύριος Γκρόκ προτείνει να συμφωνήσουμε για να συνεχιστεί η λειτουργία αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου που προωθεί την παγκόσμια ασφάλεια με την διοικητική και οικονομική βοήθεια της Ένωσης. Η προθεσμία για τροπολογίες, ε, βεβαίω ε, η μόνη δυνατή τροπολογία είναι να απορριφθεί η συνένεση, είναι το μεσημέρι της 25ης Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε εδώ 19 Νοεμβρίου και προβλέπεται να πάει στην Ολομελία του Ιανουαρίου του 17. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκάλερ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ για να δώσουμε τώρα το λόγο στους και εισηγητές. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να παρέμβει. Ε, προθεσμία... Α, δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως και εμείς θεωρούμε ότι το κέντρο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και νομίζω ότι ταιριάζει με αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα το ψήφισμα για την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών. Το ερώτημα εξακολουθεί να είναι πώς θα ε, έχουν οι λεπτομέρειες αυτού του κέντρου, αλλά αυτό μπορούμε, βεβαίως, δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εδώ πέρα, εδώ ψηφίζουμε μόνο ναι ή όχι και η απάντηση είναι σαφής πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ, υπενθυμίζω η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 25 Οκτωβρίου το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα είναι στις 29 Νοεμβρίου και θα περάσει από την Ολομέλεια τον επόμενο Γενάρη. Ε, κλείνουμε το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου. Como iba diciendo, la opinión sobre la Agencia Λοιπόν, η γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου προβλέπει 25 δεκάτου το μεσημέρι την υποβολή προθεσμίας τροπολογιών, την προθεσμία μάλλον για την υποβολή τροπολογιών. Εδώ στην Επιτροπή μας Έχουμε την πρώτη παρουσίαση της έκθεση αυτή. Η συγγετρία είναι η κυρία Μανέσκου και ο στόχο είναι να βελτιωθεί το κοινό σύστημα ασύλου. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου, ώστε να στηριχθεί, να αναπτυχθεί και να γίνει ένα φορέα που θα επιτρέπει εύρυθμα να λειτουργήσει το κοινοτικό σύστημα ασύλου. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δομικές αδυναμίες ε, του οργανισμού αυτού, αλλά επειδή δεν είναι εδώ η κυρία Μανέσκου, θα δώσω το λόγο στην κυρία Στέτινα που την αντικαθιστά. Mm. Κύριο Στέπινα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρου τη αξιότιμης συναδέλφου, της κυρίας Ρωμανέσκου, θα διαβάσω το κείμενο που μου έδωσε. Σχετικά με το σχέδιο γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την πρόταση κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου ανακαλώντας τον 439 2010 να σας πω το εξής η ε, κυρία Ραμόνα Μανέσκου σας ενημερώνει, όχι εγώ ε. στόχος της προτάσεως είναι να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστηρίξεως για το άσυλο να γίνει οργανισμός που διευκολύνει την εφαρμογή και να βελτιώσει τη λειτουργία του κοινού, του συστήματος του ευρωπαϊκού, του κοινού συστήματος ασύλου. Το Γραφείο Υποστήριξης δημιουργήθηκε το 2011 και συνεχώς υποστήριζε τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τους ισχύοντες κανόνες και να βελτιώσουν την λειτουργία των διαφόρων υφισταμένων μέσων. Η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστηρίξεω για το Άσυλο το ονομάζει Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου και μετατρέπει το φορέα αυτό σε έναν πλήρη οργανισμό, σε μια πλήρη υπηρεσία. Έτσι θα παρέχει την κατάλληλη υπηρεσιακή και τεχνική αρρωγή στα κράτη-μέλη, αυξάνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και τεχνική συνεργασία, υποστηρίζοντας την διανομή των αιτήσεων για διεθνή προστασία παρακολουθώντας και αξιολογώντας τη δυνατότητα για χορήγηση ασύλου και υποδοχή και τα διάφορα συστήματα στα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλύσουμε σωστά το κείμενο και να δούμε αν μπορούμε αποτελεσματικά να ανταποκριθούμε στις πραγματικές πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση στον τομέα της μεταναστεύσεως και του ασύλου παρέχοντας τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό συμπληρωματικά εργαλεία ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα παρόντα προβλήματα του συστήματος, κυρίως η δυσανάλογη πίεση που δέχονται τα συστήματα σύλλου και προστασίας των κρατών μελών. Έχω λάβει αρκετά σχόλια σχετικά με το κείμενο από ανεξάρτητους φορείς, ενώσεις και θα διανύμω τα σχόλια στους κοιόδης. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 25 Οκτωβρίου και η ψηφορία στην ΑΦΕΤ στις 29 Νοεμβρίου η πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Είμαι βέβαιο ότι θα υπάρξει καλή συνεργασία με τους σκιώδης εισηγητές και περιμένω αγαπητοί συνάδελφοι εσδήποτε προτάσεις ή συστάσεις έχετε όσον αφορά το κείμενο της νομοδοτήσεως. Ευχαριστώ Ραμόνα Μανέσκου. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στετίνα. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Έδειξε πω το υπάρχον σύστημα, το οποίο έχει σημαντικά ζητήματα λειτουργία, ακόμη και τι καλές περιόδους, είναι ανεφάρμοστο σε περιόδους μεγάλων προσφυγικών ροών. Το κοινό, το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου είναι ευρωπαϊκό μόνο στο όνομα, καθώς οι αρμοδιότητες και ευθύνε παραμένουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στι εθνικέ κυβερνήσει. Αν και η ενίσχυση και αυτονόμηση του οργανισμού είναι πολύ σωστό Δυστυχώ η πρόταση τη Επιτροπή δεν είναι και τόσο φιλόδοξη όσο θα επιθυμούσαμε. Αν θέλουμε να μιλάμε για ένα πραγματικά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα, τότε σήμερα θα έπρεπε να εξετάσουμε πώ ο νέο αυτό οργανισμό θα έχει την αρμοδιότητα εξέταση των αιτήσεων, των αιτήσεων ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την κατανομή του σε δεύτερο στάδιο στα κράτη-μέλη. Είναι θετικό ότι ο οργανισμό ενισχύεται με προσωπικό και δικό του υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Η δεξαμενή των 500 ειδικών από τα κράτη-μέλη, με βάση την προηγούμενη εμπειρία τη Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, είναι πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα λόγω τη συνήθι απροθυμία των κρατών μελών να παράσχουν προσωπικό στην παρούσα κρίση. Για το λόγο αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο ότι τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν ότι θα τηρήσουν τι υποσχέσει του. Σχετικά με τη διαμόρφωση του καταλόγου για τι ασφαλεί τρίτε χώρα και τι τρίτε χώρε ασφαλού διέλευση, ο οργανισμό πρέπει να έχει αποφασιστικό ρόλο και η παροχή γνωμοδότηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι υποχρεωτικό στάδιο τη διαδικασία και όχι μόνο, περίπτωση, όχι μόνο σε περίπτωση που το ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει ακόμα να διενεργεί και να δημοσιεύει ανατακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις για τις χώρες προέλευσης και τις χώρες που περιλαμβάνονται σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς καταλόγους ασφαλών τρίτων χωρών Επίσης πρέπει να δούμε να ενισχύεται ακόμη παραπάνω η δυνατότητα του οργανισμού να συνεργάζεται με τρίτες χώρες σε τομείς αρμοδιότητάς του και ιδιαίτερα στους τομείς της επανεγκατάστασης, της μετεγκατάστασης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, συμφωνώ με την εισηγήτρια στην Επιτροπή μας, αλλά και τον εισηγητή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την ανάγκη ενισχυμένη συνεργασία του οργανισμού με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, καθώς διαθέτει πλούσια εμπειρία και μπορεί να είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος. Ευχαριστώ κύριε Σοστρεβίτσιος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω εξ ονόματος του συναδέλφων του Μαριέλ Δεσσαρνές, ο οποίος μετανάστευσε και πρέπει να αναλάβω εγώ τις ευθύνες του. Λοιπόν, Σύμφωνο με την συνάδελφο ούτως ή άλλως για τα όσα μου είπε να σας μεταφέρω. Συμφωνούμε λοιπόν ότι έχει φτάσει η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να έχουν μια μακροπρόθεσμη συνεκτική στρατηγική για μια σωστή ε, πολιτική ασύλου και μετανάστευσης θα πρέπει λοιπόν να έχουν κοινή ευθύνη όσον αφορά την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων θαλασσίων και ε, στην ξηρά χερσαίων. Γι' αυτό και εγώ, η Μαριέλ δηλαδή, συμφωνούμε με την γενική κατεύθυνση της νομοθετικής πρότασης της ε, Κομισιόν μαζί με την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Ε, η Μαριέλ θέλει να τονίσει τρία σημεία τα οποία συμπλουτίσουν το κείμενο. Υπάρχει μια ανάγκη να βελτιωθεί το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης όταν μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες με την πιθανή χρήση ποσοστώσεων. Δεύτερον, μαζί με τις αντιπροσωπείες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες πρέπει να ενημερώνουμε τους δυνητικούς μετανάστες για νόμιμες διόδους και ίσως να ε, υπάρχει και ε, επεξεργασία εκεί των αιτήσεων τους. Και τρίτον, να συνδέονται καλύτερα οι χώρες διέλευσης ε, στην καταπολέμηση των διακινητών. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τους στηρίξει στην ασφάλεια των συνόρων τους και για την υποδοχή μεταναστών στις χώρες αυτές τις τρίτες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός που συζητάμε σήμερα θεωρητικά στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού για το άσυλο, ώστε να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, τόσο όταν τα εθνικά συστήματα παρουσιάζουν προβλήματα και διαρθρωτικές αδυναμίες, όσο και σε, σε καταστάσεις κρίσης. Οι εμπειρίε που έχουμε αποκομίσει τα προηγούμενα χρόνια με κάνουν να πιστεύω ακράδαντα, κύριε Πρόεδρε, πω για να γίνει βιώσιμο και αποτελεσματικό το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου χρειάζεται να γίνει καταρχήν ουσιαστικά δίκαιο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η θεμελιώδη αρχή τη δικαιοσύνη, φοβάμαι ότι πολύ απλά τόσο ο νέο κανονισμό του Δουβλίνου όσο και αυτό του ΕΑΣΟ θα καταρρεύσουν και μάλιστα αρκετά γρήγορα. Από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι θα ήταν μοιραίο λάθο αν εξετάζαμε την πρόταση αυτή μεμονωμένα, χωρίς να τις συσχετίσουμε με τις άλλες προτάσεις για το άσυλο. Όσον αφορά στον κανονισμό για τον Οργανισμό για το Άσυλο, θα ήθελα να εκφράσω τις επιφυλάξει μου σχετικά με ορισμένα σημεία για τα οποία σκοπεύω, να καταθέσω και τις σχετικές τροπολογίες άμεσα, κυρίως για το ρόλο του οργανισμού, την επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια που θα παρέχει στα κράτη-μέλη, τη συνεργασία του με τρίτες χώρες, αλλά και με την οργάνωσή του. Θεωρώ επίση απαραίτητο και θα επιδιώξω ενεργότερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι προβλεπόμενε διαδικασίε του οργανισμού, καθώ και την παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίση, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιωθεί αυτό το κείμενο. Όμω, επειδή πρόκειται για έναν κανονισμό πολύ μεγάλη σημασία που μα αφορά όλου και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα αυξημένη συγκυρία, τα χρονικά πλαίσια που τίθεται, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι ασφικτικά, όταν μάλιστα υπάρχει μπροστά μα και η Ολομέλεια. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ελπίζοντας να συμφωνήσουν σε αυτό και οι κύριοι συνάδελφοι, να προτείνω για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ευθύνες μας και να συνεισφέρουμε ουσιαστικά να δοθεί παράταση για την κατάθεση των τροπολογιών μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, μετά την Ολομέλεια, καθότι θεωρώ ότι αυτό σε τίποτα δεν επηρεάζει, αλλά αντίθετα θα έλεγα ότι διευκολύνει την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Señora Valero. Η ε, κυρία Βαλέρο, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια γενική παρατήρηση. Κάτι που είπε και η κυρία Σακοράφα. Υπάρχει πολλή νομοθεσία που βρίσκεται σε προετοιμασία και υπομελέτη για το άσυλο. Καλό θα ήταν να έχουμε λοιπόν εδώ μια στάση κάπως ε, συνεπή, κάπως συνεκτική. Διότι μπορεί να καταλήξουμε να λαμβάνουμε απόφαση για το ένα θέμα και ένα μέρος της απόφασης να αντίκειται με μια επόμενη. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε συνολικά, σφαιρικά. Και νομίζουμε ότι καλή ιδέα είναι να ενισχυθεί ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το άσυλο, έχοντα κατά νου ότι στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες. Κάποια κράτη-μέλη έχουν πολύ μακρά πείρα στην εξέταση αιτήσεων ασύλου και έχουν παράδοση στο να υποδέχονται πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ κάποιες άλλες όχι. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και μια ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας ουσιαστικά, για να έχουμε μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση στην ε, υποδοχή των ε, ετούντων άσυλων. Ιδαλώ δεν θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη ρίζα του. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι που ε, ε, να έχουν πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Και επειδή πρέπει να κάνουμε αλλαγέ, πρέπει ταυτόχρονα να βεβαιωθούμε ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται. Και πρέπει επίσης τα δικαιώματα αυτά να διασφαλίζονται. Είναι και αυτό μια ολόκληρη δουλειά. Θα πρέπει να έχει κανείς τη δυνατότητα να υποβάλει έφεση, να προβάλλει ένσταση κατά μιας απόφασης που ελήφθηκε, μιας απόρριψης έτσι σε ασύλου λόγου χάρη. Οι περισσότερες ευθύνες σημαίνουν και περισσότερη διαφάνεια. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Οι προτάσεις που βλέπουμε εδώ πραγματικά συνάδουν με το πνεύμα όσων ε, είπα και εγώ και όσων πρότεινα, αλλά θα φροντίσουμε να υποβάλουμε και κάποιε συγκεκριμένες για να ε, διευκρινιστεί το θέμα. Ευχαριστούμε. Η διαδικασία προβλέπει. Ε, δεν προβλέπει να αλλάξει δυστυχώς κάτι όπως ζήτησε η κυρία ε, Θα πρέπει λοιπόν να δεχτούμε την, ε, την ε, προθεσμία ως έχει. Θα ζητήσω τώρα την εκπρόσωπο της Επιτροπής να πάρει το λόγο. Thank you. Sorry. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια σημειώνουμε τις προτινόμενες ε, τροπολογίες ειδικά όσον αφορά την συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης και την είπατε των Θα ήθελα να αναφέρω δύο σημεία ανησυχίας. Το πρώτο αφορά την τροπολογία υπαριθμών 8 που σχετίζεται με το άρθρο 16 παράγραφος 3 σημείο G το οποίο αφορά την τεχνική αρρωγή που θα παρέχει η υπηρεσία και εκεί πέρα πρέπει να πω ότι το θέμα αυτό της βοήθειας ε, στην μετεγκατάσταση της μεταφορές είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τις συζητήσεις της ε, μεταρρύθμισης του Δουβλίνου και δεν μας αφορά εδώ. Για την τροπολογία υπαριθμών 4, το δεύτερο σημείο που ήθελα να αναφέρω, που απαιτεί πρώτερη έγκριση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και όχι μόνο της Κομισιόν όταν μιλάμε για τις ε, διευθετήσεις ε, με τρίτες χώρες. Αυτό είναι απόκληση από την κοινή προσέγγιση για τις ε, κέντρικες υπηρεσίες που έχουν εγκρίνει Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν που απαιτεί δηλαδή μόνο πρώτερη έγκριση της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με αυτό. Περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό της Σρι Λάνκα.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

appropriate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 Είναι χαρά για μας που υποδεχόμαστε εδώ την, στην Επιτροπή μας τον Πρωθυπουργό μαζί με την αντιπροσωπεία για την Νοτιοδυτική Ασία θα δώσω το λόγο στην Τζιν Λάμπερτ. Καλημέρα, ευχαριστώ που μας καλωσορίσατε. Είναι ασυνήθιστο αυτό για μένα. Που, που προεδρεύω μια συνεδριάσεως τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σας. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Το κάνω αυτό επί την ιδιότητά μου που είμαι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για την Νότιο-Ανατολική Ασία του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω εκ μέρους της Επιτροπής και της Αντιπροσωπεία τον Πρωθυπουργό τη Σρι τον κύριο Ραμίνα Κραγουασίγκα, που έχει και μαζί του και τον Υπουργό Δικαιοσύνη νομίζω, ε, νόμου και τάξης και δίπλα στον Πρωθυπουργό είναι και ο προσβευτής της Ιλάνκας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Ζοντιπαρέρα. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε μαζί μας και διάφορα μέλη του διπλωματικού σώματος για την αντιπροσωπεία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ένα θερμό καλωσόρισμα σε εσά, τον προσβευτή του Πακιστάν, των Μαλδιβών, του Μπουτάν, των Μαλδίβων και των πουτάν. Πριν δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό, να, να πω μερικά λόγια εν είδη εισαγωγής. Θεωρούμε ότι η σημερινή σα επίσκεψη αποτελεί αναγνώριση ότι η Σουηλάνκα και η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομούν ένα κλίμα εμπιστοσύνη και ένα κλίμα επαφών ως εταίροι μετά από τις περσινές εκλογές Πρέπει να πούμε δεν ήταν πάντα ομαλές οι σχέσεις όπως θα μπορούσαν να είναι, αλλά προφανώς βλέπουμε σημάδια προόδου και αυτό είναι σαφές και από τις άλλες συναντήσεις που είχατε εδώ στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα. Και οι πρόσφατες προσπάθειες για συμφιλίωση, για ε, ανανέωση οικονομική και δικαστική μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου και των συγκρούσεων που ξεκίνησαν το 2009. Όπως γνωρίζουμε όλοι η Ευρωπαϊκή Ένωση ένθερμα υποστήριζε το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευθύδια κυβέρνηση τομείς στους οποίους ε, προδεύει η κυβέρνησή σας και θα μας ενδιέφερε να ακούσουμε περί αυτών σήμερα το πρωί, διότι μάλιστα ένα σημαντικό θέμα των συζητήσεων κατά την παραμονή σας στις Βρυξέλλες είναι τα θέματα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Σρι Λάγκα. Και αυτό φαίνεται και από την εκ νέου ε, ε, αίτηση της χώρας σας για προτιμησιακό καθεστώς GSP+. Θα ξέρουν τα μέλη εδώ από το παρελθόν ότι αυτό το καθεστώς είχε απολεστεί. Δεν έγινε μια νέα αίτηση και υπήρχαν τότε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σρι Λάνκα. Ε, προφανώς οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αντικατοπτρίζονται στην αίτηση για καθεστώς GSP+. Υπάρχουν πολλές ε, προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σας. Το διαπιστώσαμε στις συναντήσεις μας και τα μέλη εδώ θα ήθελα να ακούσουν ε, το θέμα των σχέσεων ε, του πολιτικού τομέα με το στατιωτικό, κυρίως το βορρά, οι ενδοεθνοτικές εντάσεις και οι εντάσεις μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων όχι μόνο με τις μειονοτικές κοινότητες υπάρχουν προβλήματα, αλλά και με ριζοσπαστικές ομάδες και επίσης και το θέμα της ε, εκρίζωσης της ένδειας. Και λόγω της γεωγραφικής σας θέσεως μας ενδιαφέρει και η σχέση με τους γείτονές σας, όπως η Ινδία, η Κίνα και της Ενώσεως για Περιφερειακή ε, ε, Συνεργασία της Νοτιού Ασίας, ΣΑΠ. Σα καλωσορίζω εκ μέρου τη επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θέλω να πω και κάποια λόγια σαν πρόεδρο τη ε, Επιτροπή ε, για την Νοτιοανατολική Ασία. Η αντιπροσωπεία θα κάνει μια επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη στο Κολόμπο σε λίγες μέρες. Προσβλέπουμε σε αυτό. Το 2013 ήταν η προηγούμενη επίσκεψή μας. Πριν τις πρόσφατες εκλογέ θέλουμε να δούμε επιτόπου ποιες είναι οι αλλαγές και αποστολή επί δύο μέρε θα έχει διάφορε επίσημε επαφέ στο Κολόμπο και μετά θα ταξιδέψουμε να εξετάσουμε διάφορα προγράμματα στην Πατακαλώ και στην Τρικόλβη χρηματοδοτούμενα προγράμματα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, θα έχουμε την κυρία Κοχόλα και τον κύριο ε, Μαν και τον κύριο Καρίμ που είναι και ο εισηγητή στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν στην αποστολή. Θα δώσω το ε, λόγο τώρα στην εξοχότητά του τον Πρωθυπουργό για ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο και μετά θα υποβληθούν ερωτήσεις από τους παρισταμένους. Ευχαριστώ πολύ και πάλι καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Where do I begin που λέει το τραγούδι, από πού να αρχίσω. Λοιπόν, ήρθα εδώ, είχα κάλες συζητήσεις με την ύπατη εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων με την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξετάσαμε την σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σρι Λάγκα. Είχα την ευκαιρία να ξαναέρθω εδώ το 2002 όταν αναζητούσαμε μια στενότερη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σρι που περιελάμβανε την αίτηση για το μέσο γενικευμένων προτιμήσεων που κατόπιν το συνέχισε και η επόμενη κυβέρνηση του Πρόεδρου Κουμανατούγκα. Δυστυχώς οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Σρι Λάγκα ήταν τεταμένες επί τελευταίας κυβέρνησης, προηγούμενης κυβέρνησης. Οι λόγοι είναι γνωστοί και στο ζήτημα αυτό οι απόψεις του κόμματός μου ε, και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης τότε ήταν παρόμοια με της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είχαμε υποδεχθεί την τζιν στη Σρι Λάνκα, υπήρχαν άλλοι που δεν την ε, υποδέχτηκαν. Και το ερώτημα ήταν πώς θα αποκτήσουμε μια, μια δημοκρατία η οποία θα λειτουργήσει. Και τέλος πώς θα επιτύχουμε μια εθνική συμφιλίωση μετά τον πόλεμο. και να μην ξαναυπάρχουν ε, συγκρούσεις στην Σρι Λάνκα ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτικών κομμάτων στα αριστερά και στα δεξιά συναλέζει μιλ και Μουσουλμάνοι, συνδικάτα, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνία των πολιτών, για να καταλήξουν όλοι αυτοί σε μια πολιτική συμμαχία για να, για να εκλέξουμε πρόεδρο. Εκλέξαμε λοιπόν τον πρόεδρο Σίνα, ο οποίος μετά ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα. Η 19η τροπολογία του συντάγματο, μείωσε σημαντικά τις εκτελεστικές εξουσίε του πρόεδρου και επανέφερε τις ε, ανεξάρτητες επιτροπές που είχαν καταργηθεί. δικαστέ οι οποίοι είχαν ε, απομακρυνθεί χωρί να ακολουθηθούν οι συνταγματικές διαδικασίες επανήλθαν στην θέση τους ε, αλλά είπε ότι την επόμενη μέρα παρετήθηκε και είπε ότι δεν θέλω πια να αναλάβω τα καθηκοντά μου και μετά βεβαίως ορίστηκε νέος πρόεδρος του δικαστηρίου σύμφωνα με τα όσα ισχύουν. Ο Υπουργό των Εξωτερικών λοιπόν πήγε στη Γενέβη και είπαμε ας δούμε το τι θα γίνει. Και νομίζω ότι βεβαίως δεν υπάρχει εθνικός διχασμός, έχουμε και τα ΜΙΛ στην κυβέρνηση και ε, υπουργού από όλα τα κόμματα, μεταξύ των οποίων και το Τζέφνα. Βεβαίω το τρίτο κόμμα, το μεγαλύτερο, είναι η εθνική ηγεσία, η, οποία έγινε, εθνική συμμαχία η οποία έγινε ε, αξιωματική αντιπολίτευση και συνεργάστηκαν μαζί μας και αυτοί στο θέμα της εθνικής συμφιλίωσης, τα ζητήματα που αφορούν τους Ταμίλ, που αφορούν το βορρά της χώρας. Οπότε υπάρχει συντονισμός στο πολιτικό σύστημα μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΕΜΟΥ και του Προέδρου για να αποκατασταθεί η ομαλότητα στις σχέσεις ε, των εθνοτήτων στη Σρι Λάνκα. Όπως ακούσατε, έχει περάσει ο νόμος περί ελευθερίας πληροφορίας, ε, πέρασε νόμος για την υπηρεσία γνωμένων. τώρα υπάρχει μια συζήτηση για το ποιος θα πρέπει να διοριστεί εκεί πέρα. Και αυτή τη στιγμή ε, συντάσσεται ο νόμος για την Επιτροπή Εθνική Συμφιλίωση. Λοιπόν, ετοιμάζουμε επίση και νέο σύνταγμα και κοιτάμε να δούμε αν θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμό των δικαστών ε, και εξετάζουμε τη θέση των δικαστών, τη θέση των παρατηρητών και μαζί με το εκλογικό σύστημα για το πώς θα υπάρχουν ακριβώς αποκεντρωμένες εξουσίες στα επαρχιακά συμβούλια και το πώς θα, καταργηθεί, καταργηθούν οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Πρόεδρου. Ο αριθμός ατόμων που κρατούνται μειώνεται ραγδαία, όπως θα σας και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Ο στρατός της χώρας θα αποδώσει όλες τις εκτάσεις στην Τζάφνα που μπορούν να αποδεσμευτούν μέχρι το 2019. 200-300 εκτάρια είναι ακόμα υποσυζήτηση, τα υπόλοιπα θα αποδοθούν, οπότε τώρα είναι ζήτημα οικοδόμησης σπιτιών, κατοικιών τα πράγματα τα οποία συζητάμε, οι διαφωνίες είναι κυρίως το τι κτίρια θα χτίσουμε, αν θα είναι παραδοσιακά, μονόροφα, προκατασκευασμένα ή διόροφα και τριόροφα. Αυτή είναι η συζήτηση, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να συνεχίσει για πάντα. Κάποια στιγμή πρέπει να ληφθεί μια απόφαση από την Τζάφνα, από τους βουλευτές τους τοπικούς και το Επαρχιακό Συμβούλιο για να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε κάποια στιγμή. Είμαστε σε συζητήσεις για να έχουμε μια τελική συμφωνία με τη συμφωνία του Μαρτίου στην Γενέβη. και λειτουργεί και η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτά ως να σας δώσω δηλαδή μια σύντομη εισαγωγή και μετά είμαι στην διάθεσή σας και για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή αυτή. Είμαι βέβαιο ότι τα μέλη θα έχουν ερωτήσεις. Την Πέμπτη το πρωί που συνεδριάζουν οι πολιτικές ομάδες δεν έχουμε και τη μεγαλύτερη δυνατή παρουσία. Η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα μας απουσιάζει γιατί έχουν μια συνεδρίαση σε αυτή τη φάση. Ερωτήσεις. Ας, στραφούμε λοιπόν στον κύριο Καν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς σας καλωσορίζω, κύριε Πρωθυπουργέ. Χάρηκα που άκουσα αυτά που άκουσα Χαίρομαι που υπάρχει βελτίωση σχέσεων μεταξύ Σρι Λάνκα και Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είχα το προνόμιο να επισκεφθώ τη χώρα σας. Πράγματι είναι μια υπέροχη, υπέροχη χώρα. Και έχετε έξοχο πρέσβη εδώ που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Κι εγώ κατάγομαι από την Νότια Ασία. Όπως και εσείς Αγαπώ και εγώ αυτή την περιοχή. Το ΣΑΡΚ είναι πολύ σημαντική οργάνωση. Μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο εξασφαλίζοντας το ότι όλη η περιοχή θα προοδεύσει. Προχωράει ο κόσμος. Υποθέτω λοιπόν ότι έχοντας Καλέ σχέσεις η κυβέρνηση Ρελάνκα με την Ινδία και το Πακιστάν, μπορούμε να μιλήσουμε για τη διαφορά, τη διένεξη για το Κασμίρ, επί δεκαετίες υποφέρουν οι κάτοικοι του Κασμίρ. Το ΣΑΡΚ τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει, ούτω ώστε να υπάρχει σταθερότητα. Κανείς δεν θέλει να δει πόλεμο. Σίγουρα όχι μεταξύ Πακιστάν και Ινδία, που είναι και οι δύο πυρηνικές δυνάμεις. Το ΣΑΡΚ πώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί περισσότερο, να παίξει θετικότερο ρόλο για να λυθούν κάποιες από τις διαφορές και την έξι περιοχή και να ευημερήσει η όλη περιοχή. Σας ευχαριστώ. So if we collect the questions and so Mr. sorry. Yes, uh, thank you very much also once. Ευχαριστώ πολύ. Από την πλευρά μου, λέει ο κ. Γκάλερ, ε, καλώς ήρθατε. Εκτιμώ πάρα πολύ τις εξελίξεις που αναφέρατε και τις δυνατότητες για συμφιλίωση που θεωρείτε ότι υπάρχει, υπάρχουν στην περίοδο αυτή μετά τη συγκρούση. των ήμουν σχετικά νέος και σαν Γερμανός που άκουγα το BBC, το World Service, τακτικά θυμάμαι ότι τότε έλαμβα το Τρικουμβαλί, Τζάφνα, Βατικαλό, νομίζω μάθαινα τα ονόματα πόλεων από το ραδιόφωνο. Δυστυχώς, διότι ήταν αρνητικές οι περιστάσεις. Και έμαθα όμως αυτά τα ονόματα όταν ήμουν αρκετά νέος. Και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ότι τώρα αυτές οι πόλεις δεν αντιπροσωπεύουν βία, γεγονότα, επιθέσεις ή συγκρούσεις. Τούτου λεχθέντος. Η ερώτησή μου ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση όπως και του προηγουμένου συναδέλφου, αν υπάρχουν χώρες που έχουν ξεπεράσει τις εσωτερικές τους συγκρούσεις. Εν συγκρίση με Ινδία και Πακιστάν, είσαι σχετικά μικρή χώρα. Και ίσως καμιά φορά αυτό έχει σαν θετικό αποτέλεσμα ότι δεν αποτελείται απειλή για κανέναν από τους γείτονές σας, αλλά μπορείτε να είσαστε διαμεσολαβητής μεταξύ δύο μεγαλύτερων χωρών όπως είναι η Ινδία και το Πακιστάν. Ο συνάδελφος εστιάστηκε περισσότερο σε αυτό ε, τον οργανισμό το ΣΑΡΚ για την περιφερειακή συνεργασία της Νοτιού Ασίας, αλλά ίσως και διμερός ή τριμερός θα μπορούσατε ενδεχομένως να παίξετε κάποιο ρόλο, να δώσετε κάποιες συνετές συμβουλές για την αντιμετώπιση εσωτερικών συγκρούσεων, όπως ήταν το Κασμίρ που έχει και κάποια εξωτερική πτυχή το πρόβλημα. Δεν είναι αποκλειστικά εσωτερικό πρόβλημα που αφορά μόνο την Ινδία. Ευχαριστώ, λέει κυρία Λάμπερτ. Ο κύριος Αστρεβίτσιους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Χαίρομαι που σας καλωσορίζω εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων Είμαι συντονιστή ομάδων για, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, συντονιστή ομάδας μου μάλλον. Και θέλω να υποβάλω μια ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Που είναι σημαντικό τομέας. Εύχομαι να προχωρήσει καλά η Η κατάσταση μετά την σύγκρουση, μετά τι συγκρούσεις απαιτεί ε, μια σοβαρή επανεξέταση διαφόρων νόμων και έτσι να οδηγηθεί σε ένα νέο μέλλον η χώρα. Αφού τώρα η χώρα σας είναι στη διαδικασία αναδιατυπώσεως του, της νομοθεσίας της αντιτρομοκρατικής, ο νόμος αφορά συγκεκριμένα κρατούμενους και εκείνους που πέρασαν από διάφορες διαδικασίες. Η ερώτησή μου, κύριε Πρωθυπουργέ, σε ποιο βαθμό αυτός ο νόμος, ο αντιτρομοκρατικός, θα συμμορφώνεται με διεθνής τη διεθνή νομοθεσία για ανθρώπινα δικαιώματα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα ο νόμος, για να καταλάβω καλύτερα τη νομοθεσία. Η, άλλη πτυχή της ερώτησής μου. Ποια είναι η δυνατότητα να συμπεριληφθούν ανεξάρτητοι διεθνείς φορείς σε όλες τις φάσεις του μηχανισμού δικαιοσύνης και λογοδοσίας. Θα συμφωνείτε πιθανότατα ότι είναι σημαντικό νέα νομοθεσία της χώρας σας να λαμβάνει υπόψη βέλτιστες πρακτικές και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις διεθνών οργανισμών και εμπειρογνωμόνων τους ώστε να αποφευχθεί ε, τυχόν αρνητική αντίδραση ή αναποτελεσματικότητα στους νόμους αυτούς που θεσπίζει τώρα η χώρα σας. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλους τρεις. Και μετά προσθέσω κι άλλον ένα. Ο κύριος Κάλβα. Ευχαριστώ, Τζιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τη δική μου φωνή σε αυτή των συναδέλφων που σας καλωσορίσαμε σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο. Πραγματικά έχω μια ολόκληρη ε, ιστορία στο μυαλό μου από τότε που άκουσα όλες αυτές τις ιστορίες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον πατέρα μου μεγαλώνοντας ε, και είναι μια χώρα φανταστική, την έχω επισκεφτεί έκτοτε και νομίζω ότι μετά την τραγωδία των τελευταίων ετών όλοι πραγματικά ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Όμω είχα και μια μικρή επιχείρηση πέραν από το ότι ανέλαβα να γίνω βουλευτή κάποια στιγμή στη ζωή μου. Ήθελα λοιπόν να μιλήσω και για το Brexit και για το πώ πιστεύει η Σρι ότι μπορεί να επηρεαστούν οι σχέσει τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει αυτή την ε, ε, ιστορία να την κάνουμε μια ευκαιρία. Μπορείτε εσείς να το δεχτείτε έτσι, ως μια ευκαιρία που θα σας επιτρέψει ο Σρι και ως χώρα να εκμεταλλευτείτε κάποιες νέες δυνατότητες που δημιουργούνται. Δεν λέω ότι έτσι κι αλλιώς θέλουμε την αυτοκρατορία μας πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πείτε μας εσείς ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ευκαιρίες από την ε, προοπτική της κοινοπολιτείας και του Ηνωμένου Βασιλείου με την εξέλιξη του Brexit. Πιστεύετε ότι αν γίνει η όλη διαδικασία αυτή με τρόπο ομαλό μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σαφώ σε διαφορετικά στατόπεδα. Να περάσουμε στον κύριο Στέτινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Ευχαριστώ σας διαβεβαιώ ότι η σχέση μου με τη χώρα σας είναι εντελώς προσωπική. Θαυμάζω από παλιά τη Σρι Λάνκα. Δυστυχώς τελευταία φορά βέβαια ήρθα πριν από πολλά χρόνια. Και βρέθηκα στη χώρα τη στιγμή που οι εχθροπραξίες με τους Ταμίλ ήταν ε, στο Ζενίθ. Τώρα, για τις εθνοτικές μειονότητες, τι λύση έχετε βρει. Μάλιστα, ευχαριστούμε ο κύριος Φρέντ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ήθελα να έχουμε μία κόντρα με τον κύριο Γκάλερ, αλλά δυστυχώς έφυγε. Δηλαδή, η δική μου ανάμνηση του τι συνέβη τότε, αφορά μια από τις προ-προ-προκατόπουσες, την κυρία Μαντεραμάνκε, η οποία από το 60 έως 65 και από το 70 έως το 77 είχε την Πρωθυπουργία και όταν σκέφτομαι τι άκουσα, σκέφτομαι τον πόλεμο τότε, σκέφτομαι και τον πόλεμο του Βιετνάμ και πόλεις ε, σαν την Ουέι και το Chi Μια από τις καλύτερες φίλες μου πάντως είναι μια κυρία από τη Φιλάγκα η οποία από τη Βιέννη τώρα έχει φτάσει να ζει στη Νέα Υόρκη. Και έχουμε πολύ στενή προσωπική σχέση και με την ίδια και με την οικογένειά της. Όμως αυτά που θέλω να σας ρωτήσω είναι διαφορετικά. Γιατί περάσατε ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο στη χώρα σας. Και με συγχωρείτε που καθυστέρησα κάπως γιατί δεν άκουσα τα πρώτα 2-3 λεπτά της ομιλίας σας. Πιστεύετε ότι αυτός ο φρικτός πόλεμος έχει πραγματικά αυτή τη στιγμή ε, πάυσει και συγκρατείται, συγκρατούνται οι δύο πλευρές ή μπορεί να προκύψουν σπίθες και να υπάρξει αναζωπήρωση. Μήπως τα πράγματα απλώς τα έχουμε σπρώξει κατά το χαλί ή μπορεί να ξαναξεκινήσει η κόντρα. Δεν ξέρω πολλά ε, για το θέμα. Ίσως να μας λέγατε εσείς πώς το βλέπετε το θέμα τώρα. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να προσθέσω μια ερώτηση. Για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με την οικονομία. Τα μέτρα που προβλέπετε για την καταπολέμηση της φτώχειας. Όταν ήρθαμε τελευταία φορά στη Σιλάνκα, μια από τις περιοχέ που επισκεφτήκαμε ήταν οι θητείε τεϊόδεντρων. Και είδαμε ότι για τους ε, εργαζόμενους εκεί οι συνθήκες ήταν πραγματικά πολύ χαμηλού βιωτικού επίπεδου, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα ε, χρειάζεται προγνωσμένη ανάπτυξη. Πώς το βλέπετε λοιπόν αυτό, πώς θα μπορούσε να αλλάξει. Πάντως, ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις. Μιλήσαμε για το ΣΑΡΚ, για τον εμφύλιο πόλεμο, για τον νόμο κατά της θερμοκρατίας. Ήταν ερωτήσεις που εγώ ήθελα να θέσω. Το αν αυτή η αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή έχει οριοθετηθεί και τι σχέση θα αναπτύξετε ε, με την κοινοπολιτεία ε, διότι με τον προηγούμενο πρόεδρο η συνεργασία δεν είναι πάντοτε αγαστή στα πλαίσια της τοπικής κυβέρνησης και τη κοινοπολιτεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσει. Το Κασμίρ είναι μια ε, σύγκρουση μεταξύ δύο διαφορετικών πλευρών. Δεν μπορεί να συγκριθεί ακριβώ. με το Σάρικο. Όμως, εκεί που βρισκόμαστε εμείς, θα μπορούσα να, να σκεφτούμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητούν στις συναντήσεις τους στο Κασμίρ. Θα μπορούσαν να φέρουν μαζί τους ηγέτες του Πακιστάν και τη Ινδία για να έχουν συνομιλίες. Όμως, το ΣΑΡΤ στόχο έχει να φέρει μαζί τους δύο ηγέτες για να συνομιλήσουν, αλλά και για να προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία σε άλλα ζητήματα, την παιδεία, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, σε πολλούς άλλους τομείς, ώστε να αμβληνθούν οι σχέσεις, οι οξύες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο πολλά από αυτά έπαψαν να προχωρούν. Και φτάσαμε σε μια κατάσταση παρόμοια το Κασμίρ. Τελευταία σύνοδος μάλιστα δεν μπορέσε καν να διοργανωθεί. Μετά την ε, επίθεση στο Κασμίρ και τη δυσυνοριακή τρομοκρατία. Οπότε, ε, εφόσον ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούν να πάρουν μέρος στα, στις συναντήσεις του ΣΑΡΚ, το όλο θέμα αναβλήθηκε. Το Κασμίρ λοιπόν είναι ένα θέμα διμερές, αλλά τελικά οδήγησε σε κατάρρευση και τις όλες της ΣΑΡΚ. Θα πρέπει οι δύο κυβερνήσεις μεταξύ τους να βρουν μια λύση. Εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χαλαρώσουν τα πράγματα, αλλά θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ καιρό όλο αυτό. δεν μπορεί να επιληθεί αν δεν συναντηθούν οι δύο πλευρέ. Οπότε αυτός που θα την πληρώσει θα είναι το ΣΑΡΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς περιέχουν τα, οι επιστολές που αποστήλαμε. Αλλά υπάρχει και η συνόδος του BIMSTEC που είναι προγραμματισμένη Τώρα άμεσα Ινδία, Σιλάνκα, Μπαγκλαντές, Μιανμάρ και Ταϊλάνδη. Ένα πενταμερές σύστημα, ε, μάλλον, ε. ε, έχουν σύνοδο την ίδια ώρα με τις BRICS, ε, τις χώρες BRICS Δεν είναι γνωστό ακόμα πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν οι ατζέντε αυτών των συναντήσεων. Δεν, σας, δεν θα σας πω ακριβώς λοιπόν τι πρόκειται να συζητήσουμε, αλλά ανησυχούμε. Ανησυχούμε για το πώς θα εξακολουθήσει το ΣΑΡΚ. Δεν βλέπω να γίνεται πόλεμος προς στιγμή. Σίγουρα δεν θα γίνει πόλεμος. Η ειδική πλευρά όμως επιμένει να ληφθούν ισχυρά μέτρα. Για τη διασυνοριακή τρομοκρατία Να δούμε λοιπόν πώς θα προσεγγίσουμε το όλο θέμα και αν δεν πετύχουμε να πω ότι το μέλλον του ΣΑΡΚ σίγουρα απειλείται. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα ευρύτερο. Δεν μπορώ εγώ να παραποφάσω να το σχολιάσω περαιτέρω. Επόμενο εάν θα υπάρχει άλλος, αν θα γίνει πάλι πόλεμο στη Σρι Λάγκα. Η απάντησή μου είναι όχι. Ο εμφύλιος τελείωσε. Είναι πολλά τα μέτρα που λάβαμε σε σχέση με τις εθνοτικές μειονότητες Και το θέμα είναι βέβαια να υπάρξει και οριστική συμφιλίωση. Έχουμε περάσει συντακτική συνέλευση για να συνταχθεί ένα νέο, για να υπάρξει ένα νέο σύνταγμα. Το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με αυτό και ο κοινοβουλευτισμό μα. Είναι κάτι το οποίο όλοι το θέλουμε με περαιτέρω ε, εκχώρηση αρμοδιοτήτων στι περιφερειακέ αρχέ. Όχι λόγω κομματικών ε, προτεραιοτήτων, αλλά του τι ζητήματα είναι τα πιο επίγοντα. Με περισσότερες, λιγότερες προτεραιότητες, ε, μακρύ και πιο περιορισμένου καταλόγου και έχουμε φροντίσει ε, κάποιοι από τους βασικούς υπουργούς και κάποια από τα μέλη της κυβέρνησης να ε, επι, μπορέσουν αυτές τις προτεραιότητες που είχαν να τις κάνουν να ακουστούν. Περισσότερη εκχώρηση εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. Ένα άλλο θέμα είναι η ανάγκη να δημιουργηθεί γερουσία. Εδώ μπορεί και να υπάρχει πρόβλημα διότι γίνεται αποδεκτή ανάγκη για γερουσία από την EMA, αλλά η Λάγκα δεν διαφέρει από τις άλλες χώρες. Δεν είναι πολύ ευχάριστο να προσθεθεί κι άλλο ένα σώμα εκλεγμένων και με πέντε μέλη ανά επαρχία. Τέλος θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Αυτό που λέμε είναι κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο να εκλέξει πέντε μέλη για την Γερουσία. Και να είναι και άλλοι και όχι μόνο υπουργοί. Δεν ε, θα προβλέψουμε περισσότερα πόστα όμως, απλώς θα πρέπει να κοιτάξουμε να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί στο Κολόμπο. θα δούμε λοιπόν πόσοι θα είναι το κοινοβούλιο την άλλη θα προκρίνει 8 εξέφρες προσωπικότητες για να έχει 55 μέλη γερουσία και τα μέλη της γερουσίας θα έχουν τη δυνατότητα να αναπέμψουν νομοθετικές πράξεις στο Κοινοβούλιο για να τα ξαναδούν. Αλλά και το Κοινοβούλιο όταν πρέπει να εγκρίνει κάποια, κάποια νομοθεσία για συγκεκριμένα θέματα ε, θα υπάρχει η ίση μεταχείριση και από τις δύο πλευρές. Για την ώρα αυτό που κοιτάζουμε είναι ότι οργανώνουμε τα δύο σώματα, ε, διοργανώνουμε τα ίδια τα κτίρια όπου θα στεγαστούν, τα κοινοβούλια και τελικά ε, τα μέγαρα αυτά είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι προηγουμένω, γιατί είχαν ισοπεδωθεί τελείω. Υπάρχει πάντω ε, τεράστια προσπάθεια ήδη με την λεγαόντωση να φτάνει σε περιοχέ που δεν υπήρχε ποτέ. Η κοινωνική δυσκολία που υπήρχε προηγουμένω δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι κάποιοι δεν έχουν όλη την οικογένεια κοντά του. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν μεταναστεύσει και μπορεί να έχει κρατήσει πολύ ο πόλεμο και τρει-τέσσερι γενιέ προηγούμενε να έχουν πολλά μέλη που του λείπουν, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό διαρκώ ανανεώνεται. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο λοιπόν για να αναμοδιαφερθεί ο κοινωνικό ιστό. Και κάτι άλλο που είναι αλληλένδετο με όλα αυτά είναι ότι ο κόσμο παίρνει εμβάσματα από του συγγενεί στο εξωτερικό, δεν λένε όχι. Όμως μερικοί τα χρησιμοποιούν αυτά μόνο και μόνο για να τα πιούνε και να πάρουν ναρκωτικά. Έχουμε πρόβλημα προβληματισμό στα ναρκωτικά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Είναι αυτό προφανώς ένα πρόβλημα για τους κυβερνώντες. Αλλά το άλλο πρόβλημα είναι η μετακίνηση του πληθυσμού εσωτερικά. Δηλαδή είναι πολλοί αυτοί που έχουν έρθει να μένουν στο Κολόμπο. Πώ θα του πάμε πίσω στι περιοχέ του, Αυτό είναι ένα ερώτημα. Κοιτάζουμε εάν μπορούμε να του δώσουμε τα κίνητρα για να πάνε να. <coughs> να επενδύσουν στις περιοχές από όπου έρχονται. Τζέφνα λόγου χάρη. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε να μας βοηθήσουν να ετοιμάσουμε ένα πακέτο για το Βορρά και την Ανατολή ή το Βορρά. Θέλουμε επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε σε εσά ή θα θέλαμε να έρθετε, να δείτε την κατάσταση. Χρειάζεται ένα ξεχωριστό πακέτο για την Τζαφνά. πρέπει να αποπληρώσουμε και τα δάνεια που έχουν αναλυφθεί από το προηγούμενο καθεστώ. Συντονιζόμαστε με το δούνο του, αλλά πρέπει όμω να βοηθηθούμε και απ' έξω για να προχωρήσει η οικονομία σε τσεφνά. Όταν έχουν χρήματα οι άνθρωποι, χτίζουν σπίτια, προχωρά η οικονομία. Αυτό ζητάμε, ε, ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια δολάρια, ούτω ώστε να κινηθεί η τσέφνα. Και ζητάω τη βοήθεια και, της, ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι έχετε δύσκολες, ε, δύσκολους οικονομικούς περιορισμούς, αλλά αν δοθεί αυτή η βοήθεια θα λυθούν τα προβλήματα, άπαξ διαπάντως. Μετά, ανθρώπινα δικαιώματα. Ετέθησαν δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Συζητούμε τον κανόνα των παρατηρητών στα δικαστήρια. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Κυρίως σε ειδικά δικαστήρια. Όχι απλά δικαστήρια, σε ειδικέ υποθέσεις. Αν έρθουν οι παρατηρητές, τι δικαιώματα έχουν, τι έγγραφα μπορούν να ζητήσουν. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να παρακολουθήσει τη δίκη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα δικαιώματα των παρατηρητών θα πρέπει να καθοριστούν και είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητούνται. Τώρα, όσον αφορά τον αντιτρομοκρατικό νόμο, έχουμε το νόμο για την περιφερειακή ε, τρομοκρατία. Αντιγράψαμε την νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου του 1974 και κάναμε τροποποίησεις μέσω του κανονισμού για τη δημόσια τάξη, των διαφόρων ρυθμίσεων για τη δημόσια τάξη και χρησιμοποιήθηκε και για ανθρώπους που κρατούνται. Δεν έχουμε κρατουμένους σε αυτή την κατηγορία τώρα, διόριστα ε, μία επιτροπή να εξετάσει την νέα νομοθεσία. Έχουν υπογράψει στην έκθεση τα 17 εμπλεκόμενα μέρη, 17 εμπλεκόμενοι φορείς. Έχουμε ετοιμάσει μία λευκή βίβλο, θα εξεταστεί από την αρμόδια ελεγκτική επιτροπή και θα στείλει στους άλλους αρμόδιους φορείς το έγγραφο αυτό. Αυτή η λευκή βίβλος δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα, εμπεριέχει συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής. Θα γίνουν κάποιες τροποποίησεις. Ο Υπουργός ή εμπειρογνώμων του ΟΗΕ θα μπορούσαν να αναφερθούν σε αυτό. Πολλές χώρες θέλαν να μας βοηθήσουν με την όλη διαδικασία. Ζητήσαμε η βοήθεια αυτή να διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών και της διευθύνσεως της εκτελεστικής της αντιτρομοκρατικής του ΟΗΕ. Έχουμε ετοιμάσει τις προδιαγραφές. Η Λευκή Βίβλος συζητείται μέσω των ελεκτική, της Ελεκτικής Επιτροπής αλλά και το προσωπικό του ΟΗΕ θα κάνει τα δέοντα. Θα έρθει σε επαφή με τις ε, ε, Ελεκτικές επιτροπές και την κοινωνία των πολιτών. Όσον αφορά τους κρατούμενους, Έχουμε πέντε κρατούμενους οι οποίοι θα απελευθερωθούν μέχρι το τέλος ε, του μηνός. Θα, δεν θα έχουμε κανέναν μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 41 είναι σε προσωρινή κράτηση και περιμένουν την απαγγελία καταγγελιών και την ε, κίνηση ποινικών διαδικασιών. Και άλλους 11 έχουν τελειώσει οι ποινικέ ε, έρευνες και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. 96 εντάλματα ε, συλλήψεως υπάρχουν στο νότο δικαστήριο. Συμπεριλαμβάνονται εκεί αυτοί αυτούς που έχουν αθωωθεί αν θέλετε ή τους έχει δοθεί χάρη. Με τη νέα κυβέρνηση κάναμε διαδικασία και εκείνοι μπορούσαν να απελευθερωθούν με πολύ μικρές κατηγορίες απελευθερώθηκαν. Σε άλλους προσφέραμε τη δυνατότητα αποκατάστασης. Ε, δεν ήθελαν να κάνουν κάτι να, να τους πάμε σε κέντρα αποκατάστασης αν θέλετε και θέλανε να περάσουν από τη δίκη μέσω σοφρονιστικών διαδικασιών και θα να πέσουν από δίκη. Εκείνοι που πέρασαν μεγάλο χρονικό διάστημα σε προσωρινή κράτηση και ίσως τελικά η προσωρινή του κράτηση ε, κράτησε περισσότερο από ότι αν είχαν καταδικαστεί κανονικά για το διαπραχθένα δίκημα. Θα εξεταστούν όλα αυτά. Νομίζω πως όταν θα έρθετε στο Κολόμπο με την αντιπροσωπεία θα συναντηθείτε και με τις ομάδες άνθρωπινων δικαιωμάτων. Τώρα για την οικονομία. Υπάρχει μια ύφεση. Κοιτάξτε, δεν ε, υπήρχε όφελος για τον λαό μετά το τέλος του πολέμου ακόμα. πρόθεσμα λοιπόν το 2015 στόχο έχουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αυξηθεί. Η ζήτηση αυξήθηκε αλλά υπήρχε βεβαίως και πληθωρισμός. Και υπήρχαν και αυξήσεις στους μισθούς και τα λοιπά. Τώρα έχουμε μια οικονομία την οποία ε, το... Η... Η συλλογή των φόρων ε, ήταν ε, γύρω στο 11% του ΑΕΠ. Υπό τον προηγούμενο Πρωθυπουργό ήταν 70%. Οπότε έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Οι εξαγωγές επίσης έπεσαν ε, και υπήρχε και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, γιατί είπε η κυβέρνηση ότι δεν θέλουμε σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και προτιμούσαν να στέλνουν κόσμο να δουλεύει στη Μέση Ανατολή για 300 δολάρια το μήνα. Και χάσαμε την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών μας. Και οι τουρίστες επίσης βεβαίως. Το πρόγραμμά μας τώρα είναι ακριβώς να προωθηθεί αυτό. Και η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ σημαντική. Οφείλω να πω ότι κάναμε τις διαπραγματεύσεις έχει αρθεί η απαγόρευση αλίας, οπότε τώρα μπορούν να δουλέψουν οι ψαράδες. Υπάρχει περισσότερος τόνος στην ευρωπαϊκή αγορά και στις, ε, κουζίνες των ανθρώπων. Ψάρι. Προσπαθούμε, όπως σας είπα, να γίνουμε ανταγωνιστικοί με την κινέζικη αγορά, με την αγορά της Σιγκαπούρης, την Ινδική αγορά και αυτά είναι τα προγράμματα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας δρόμος που κατασκευάζεται, μια κινέζικη πρωτοβουλία. Φτιάχνουμε και έναν κόμπο το Αμπάτο Ντεάσι σε μια πολύ φτωχή περιοχή. Και όπως αναπτύσσονται αυτά, οπωσδήποτε θα βοηθήσει τη βιομηχανία, των τουρισμών στις στοχές αυτές τις περιοχές ε, και από τις φοιτίες ο κόσμος θα πάει εκεί να γίνει εργάτης. Επίσης και οι βιομηχανίες ε, φεύγουν ε, από τις δυτικές περιφέρειες και αναπτύσσονται και μέσω μακροπρόθεσμα σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και την περιοχή του λιμανιού Κρυμκολή και η ανατολική και η νότια περιοχή και η ενδοχώρα θα γνωρίσει αύξηση του τουρισμού. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά. Η μεταρρύθμιση βεβαίως ε, της γεωργίας θα χρειαστεί περισσότερο. Το καουτσούκ έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή και οι τιμές του τικ έχουν πέσει δεν είναι σε καλή κατάσταση οι φοιτίες, χρειάζονται αναδιάρθρωση. Αυτό το οποίο κάναμε λοιπόν είναι ότι ε, δίνουμε γη και χρήματα για να μπορέσει ο κόσμος να χτίσει σπίτια ε, σε ακτήμονες. Τους δίνουμε λοιπόν αγροτεμάχια και σταδιακά θα χτιστούν 30.000 ε, σπίτια τα επόμενα 4-5 χρόνια και κάποιοι ίσως φύγουν. Το ζήτημα λοιπόν είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε εκεί και αν θα μπορέσουν να έχουν βεβαίως ε, και τις κατάλληλες τιμές του τσαγιού. Γιατί και οι πιο εκπαιδευμένοι φεύγουν από την Ήπεθρο σε όλες τις φοιτίες υπάρχουν δύο μόνο ε, σχολές ε, με σχετικές επιστήμες, γεωπονικές και τέτοια. Οπότε θα ξεκινήσει και αυτός ο κλάδος μετά. Κάναμε την υποχρεωτική εκπαίδευση 13 χρόνια. Για να μένει ο κόσμος στο σχολείο. Και Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα μοιράσουμε τάμπλετ και οι φοιτητέ θα παίρνουν ε, δάνεια με πολύ ευνοϊκού όρου για να αγοράσουν λάπτοπ. Υπάρχει όπω είπα και έλλειψη στέγη. Και υπάρχει βεβαίω και το πρόγραμμα εκμάθηση αγγλικών όσον αφορά την ιδιοκτησία τη γη. Όπω ξέρετε, εδώ και γύρω από τη δεκαετία του 1930 δίνονταν γη σε μικροκαλλιεργητές με δάνειο από το κράτο, ω δάνειο από το κράτο. Δηλαδή η γη ανήκε στο κράτος και απλά εμπιστονόταν. Αλλά τώρα θα παίρνουν τίτλο ιδιοκτησίας της ε, γης. Εκατομμύρια άνθρωποι. Με έγγραφα τα οποία βεβαίως μετά θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν κι άλλο. Και στοχεύουμε ιδιαίτερα τις ε, φτωχές περιοχές και θα υπάρξει κάποια κινητικότητα. Οι πιο ικανοί θα φύγουν ίσως από τα χωριά, αλλά κινητοποιούμε ακριβώς την οικονομία της υπαίθρου για να μην υπάρξει κατάρρευση. Και βεβαίω βλέπουμε και κάποια αυξημένη παραγωγικότητα. Μετά υπήρχε ένα ερώτημα για την κοινοπολιτεία και το τι μπορεί να γίνει. Ε, κοιτάξτε, 47% των εξαγωγών μας πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανησυχούμε το τι θα γίνει όταν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μηνύματα από την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι τόσο καλά. Ελπίζουμε να μην ε, πέσει ή μειωθεί πάρα πολύ γρήγορα γιατί Εμείς στοχεύουμε κυρίως στις αγορές χαμηλότερου εισοδήματος. Ενδύματα φτηνά, και τσάι. Οπότε μπορεί να μας επηρεάσει αυτό. Καλωσορίζουμε όμως τις επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί ε, αν φύγουν από την Ένωση θα πρέπει να επενδύσουν κάπου αλλού. Μετά το άλλο θέμα είναι αυτό το οποίο είπαμε σε μια συνάντηση στο Κολόμπο. Η ανάγκη να υπάρχουν στενότερες σχέσεις ε, εμπορίου και επενδύσεων. Και το είχαμε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, τον ε, Τζον Κίθ, πώς θα έχουμε μια συμφωνία στο πλαίσιο της κοινοπολιτείας για εμπόριο και επενδύσεις. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις ε, τεθεί σε ισχύ το άρθρο 50 και βεβαίως υπάρχουν οι περιορισμοί γιατί υπάρχουν πολλές χώρες ε, και το θέμα είναι το τι θα κάνει η Ινδία, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, οι μεγάλες αφρικανικές χώρες. Ίσως η Ινδία θα μπορούσε να στείλει κάποιους ειδικού ε, και αναμένουμε τα αποτελέσματά τους βεβαίω. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο επί καιρών εστιαζόταν σε ένα άλλο σύστημα, όχι στο εμπόριο. Π.χ. η Αυστραλία η Νέα Ζηλανδία κάνουν εμπόριο με την Κίνα. Η Ινδία έχει δική της αγορά. Ανατολική Αφρική είναι διαφορετική από τη Δυτική Αφρική. Η Καραϊβική το ίδιο. Οι Καναδοί προσπαθούν να διαπραγματευτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπωσδήποτε, ναι, θα είναι κάτι το μακροπρόθεσμο, δεν είναι βραχυπρόθεσμο και εμείς πρέπει να μελετήσουμε Βεβαίω το θέμα είναι όντω και τι θα γίνει πέρα με την Σιγκαπούρη. Περισσότερες από αυτές τι χώρες είναι στη Βρετανική κοινοπολιτεία και έχουν μια Βρετανική επιρροή. Οπότε εξετάζουμε κάποιες ε, χωριστέ ε, διευθετήσεις. Και σε ελπίσουμε ότι διάφοροι υψηλόβαθμοι άνθρωποι θα τα μελετήσουν αυτά και θα μπορέσουν να επανέλθουν, αλλά δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε εκ βαθέων, Πρωθυπουργέ, για αυτές τις τόσο διεξοδικές σας απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολλά από αυτά που μας είπατε, το τι θα γίνει στο μέλλον, οι εμπορικές διευθετήσεις Και βεβαίω όσοι συμμετέχουμε στη μεικτή κοινοβουλευτική αλλά και όλοι οι συνάδελφοι στο Ευρωκοινοβούλιο ενδιαφέρονται να δούνε ακριβώ την ε, ε, συνέχεια των ε, εξελίξεων όλος ιδιαίτερα στο κοινοβούλιο μας. Περιμένουμε να δούμε ότι οι αλλαγές που γίνονται όντως θα ριζώσουν και ότι ο πόλεμος πραγματικά έχει λήξει. Αυτό θα είναι ε, προς όφελος όλων των πλευρών στην ε, Σρι και είναι κάτι που θέλουμε να ε, ολοκληρωθεί. αυτή την πολύ θετική εξέλιξη που να κρατήσει για πολύ καιρό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Υπουργό Εσωτερικών που ήρθε εδώ Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση του συναδέλφου από τους φιλελεύθερους που θα δεχτείτε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ που δεχτήκατε, κυρία Τζιν Λάμπερ, να πέτρεψε αυτό το μέρος της συνεδρίασης. 24 ε, ε, Οκτωβρίου, τη Δευτέρα στο Στρασβούργο είναι η επόμενη συνεδρίασή μας, με τις ψηφοφορίες και μετά στις 28 στις 7 και 8 Νοεμβρίου, μάλλον στις